Μετά έχουμε το θέμα της Συρίας, ε, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιες πάλι ευάλωτες κοινότητες. Μπίελαν λοιπόν από τους συντάκτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν φαίνεται ακόμη βελτίωση της κατάστασης στη Συρία και η συνεχόμενη σύραξη ε, κόστισε τη ζωή σε 150.000 ε, άτομα. Επίσης έχουμε ε, σχεδόν αποδείξει για τη χρήση χημικών όπλων κατά του άμαχο πληθυσμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τη Συρία. Θα πρέπει όμως κατηγορηματικά να ζητήσουμε αποχώρηση του Μπασαράσαντ από, το, από την κυβέρνηση. Έχουμε όλο και συχνότερες περιπτώσεις δίωξης χριστιανών. Μόνο πέρυσι 1.200 ε, άτομα της χριστιανικής μειονότητας έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα με χρηματοδότηση τσιχαντιστών και τρομοκρατικών οργανώσεων μπροστά στα μάτια της, ε, ε, της κυβέρνησης στο Χαλέπι, στη Χόμς, εξολοθρεύτηκαν μεγάλες θρησκευτικέ χριστιανικές κοινότητες. Θα πρέπει να καταδικάσουμε την Συριακή κυβέρνηση και κυρίως τις βαναυσότητες και τις επιθέσεις κατά των χριστιανών. Δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα αυτά τα εγκλήματα. Θα πρέπει να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την αιματοχυσία. Και μάλιστα οι διπλωματικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν κέρια σημασία, γιατί η Αγγής Ανατολή είναι ε, γειτονική περιοχή. Θα πρέπει ε, να βοηθήσουμε λοιπόν τους ε, Σύρους ε, πολίτες όπως και τους συμμάχους μας που, όπως η Τουρκία. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στην παγκόσμια κοινότητα προκειμένου να διορθωθούν αυτές οι επονίδιστες διώξεις και διακρίσεις και να σταματήσει αυτή η αδικαιολόγητη σύραξη. Λυπούμε για την δολοφονία του ιερωμένου Βαντερλούχτ που από αλληλεγγύη προς τους κατοίκους της πόλης Χόμς έμεινε στην πολιορκημένη πόλη χάνοντας τη ζωή του. Θα πρέπει ανεξάρτητος δικαστής ε, να ασκήσει δίωξη κατά των δραστών αυτής της στιγμής δολοφονίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά ο κύριος Πέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πάτερ Φραντς Φαντερλούχτ έφυγε από κοντά μας, έφυγε από τους πολιορκημένους της Χόμς, από τις χριστιανικές κοινότητες. Δολοφονήθηκε φρικτά. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια. Κυρίως για το μέλλον της Συρίας του, αλλά και για εμάς εδώ πέρα, στην Ευρώπη. Γιατί ο Πάτερ Φαντερλούχτ, ο Πατήρ Φαντερλούχτ, ήταν πραγματικά μια μορφή η οποία μαχόταν για την ειρήνη ενάντια στον σατανικό σαλαφισμό. Και εδώ πέρα φταίνε και πρέπει να ντρέπονται και οι Ευρωπαίοι τζιχαντιστές. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και υπάρχει και άλλη μια παράληψη στο ψήφισμα. Δεν λέει τι έγινε στην και ΣΑΠ τον προηγούμενο μήνα χριστιανικό μέρος στο οποίο επιτέθηκαν οι τζιχαντιστές. Μιλάει βεβαίως για τις επιθέσεις των Τούρκων. Και βεβαίως πρόκειται για τους απογόνους αυτών που γλίτωσαν από τη γενοκτονία του 95-96. Πρόκειται για Ισλαμιστική επίθεση κατά των χριστιανών του Κεσάπ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μετά από όλα αυτά να μιλάμε σοβαρά για το ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα και να μην σπάμε το ταμπού που υπάρχει σχετικά με την Άγκυρα. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα τιμάμε τους χριστιανούς μάρτυρες των πατέρα Φαντερλούκτ μεταξύ αυτών, αλλά και τα αμέτρητα θύματα όλων των θρησκειών και ομολογιών που έχουν πεθάνει μέχρι στιγμή στην Συρία. Υπάρχουν λοιπόν δύο τεράστιες μιλόπετρες. Από τη μία έχουμε το καθστός Άσαντ, από την άλλη τους τζιχαντιστές που πραγματικά θέλουν να κάνουν ένα φανατικό θεοκρατικό κράτος και ανάμεσα σε αυτές δύο μιλόπετρες κινδυνεύουν να αφανιστούν οι μειονότητες της Συρίας μεταξύ των οποίων και οι χριστιανοί. Αν θα παρέμβουμε εμείς ως Ευρωπαίοι για να μεσολαβήσουμε και να συνομιλήσουμε με τα κομμάτια εκείνα της αντιπολίτευσης που δεν θέλουν να επιβάλλουν αμία άλλη τυραννία δεν θα το κάνει κανείς και πρέπει να μιλήσουμε και με τα κομμάτια εκείνα του καθεστώτος που θέλουν ειρήνη. Και πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Δεκαϊζερ για την καλή συνεργασία που εμφανίζεται και σε αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Για τρία μισή λεπτά η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η τέταρτη φορά που θα ψηφίσουμε κάτι που αφορά τη Συρία απέτυχαν οι διαπραγματεύσει Γενέβη 2, υπάρχει κατακαιρματισμό τη απόψη και οι θρομοκρατικέ επιθέσει αλλά και η αδιαφορία του καθεστώτο οδηγούν ε, σε αυτό το τέλμα όπου ένα ακόμη ψήφισμα δεν θα αλλάξει τίποτα για τον πληθυσμό και του πολίτε τη Συρία. Αλλά το ψήφισμα αυτό το θέλουμε παρόλα αυτά. Διότι τίποτα δεν είναι χειρότερο από τη σιωπή σε αυτέ τι περιπτώσει από την πλευρά τη διεθνή κοινότητα. Ε, θελήσαμε πρώτα απ' όλα το ψήφισμα αυτό για να αποφύγουμε το θάνατο γυναικών και ανδρών των οποίων η δέσμευση και αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, ανεκτικότητα και την προστασία τη ελευθερία τη έκφραση και των συνειδήσεων είναι κάτι το αναντήρητο. Θα πρέπει η κυρία Τουνέ που ήταν, ε, ε, Σατουνέχ που ήταν ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και σήμερα έχει απαχθεί με τον σύζυγό τη και του συγγενεί τη να βρεθεί. Θα πρέπει ο πατήρ Πάολο που τον γνώρισα και εγώ στην Συρία το 2008 όταν ήρθε μαζί με την κυρία ε, Σαραζάντ στην ε, Ευρώπη για να ζητήσει βοήθεια εκ μέρου των Σύρων, θα πρέπει και για αυτού να γίνει κάτι. Ο πατήρ Φαντελούχ που έμεινε κοντά στου χριστιανού και του μουσουλμάνου τη Χόμ χωρί να κάνει διακρίσει, ήταν και εκείνο ένα άνθρωπο που πέθανε στον ίδιο γόνα στο πλευρό μα. Ε, πίσω από εμά βρίσκονται άνδρε και γυναίκε, εκατοντάδε, εξαιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή του για την ελπίδα, τη δημοκρατία, την ελευθερία και για Στι πρώτε τάξει ε, τη επανάσταση του 2011. Δεν πρέπει να του προδώσουμε και δεν θα πρέπει να του αφήσουμε να υποφέρουν στη σιωπή ε, μαζί με τον τοπικό πληθυσμό. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να αναλάβουμε δράση γιατί έχουμε δύο πρόσφατα φαινόμενα. Το πρώτο που έχει να κάνει με τη συγκρούση και τι ε, θανατικέ καταδίκε που σήμερα πλήττουν τι θρησκευτικέ μειονότητε και που υποδαβλίζονται από το καθεστώ, αλλά και τι εξωτερικέ επιδράσει που βαρύνουν ιδιαίτερω αυτόν τον ε, δανεικό, τον ε, εικονικό πόλεμο. Θα ήταν λοιπόν αρνητική στάση εκ μέρους μας, θα ήταν άρνηση πλήρως να ε, μην δούμε ότι στην ε, Μαλούλα αυτά που συνέβησαν ήταν ουσιαστικά μια ανατροπή της επανάστασης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους, τις οικογένειες των θυμάτων και να ακούσουμε τις μαρτυρίες όσων δέχτηκαν επίθεση, όσων υπήρξαν θύματα καταδίκη ε, καταδίκης και εκτέλεσης. Θα πρέπει να δούμε τι έγινε στην περίπτωση της Χόμς, αλλά και που μιλάνε ακόμα αραμαϊκά ή τι γίνεται στην αρμενιακή πόλη της ε, Κεσάμπ όπου δεν υπήρξαν μόνο στρατιωτικές ε, παρεμβάσει, αλλά και έχουμε και χριστιανικές μειονότητε που πρέπει να προστατευτούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και το δεύτερο φαινόμενο που είναι θλιβερό με την παρουσία τρομοκρατικών ομάδων οι οποίε είναι παρούσες, χρηματοδοτούνται τους ε, εγκληματίες τζιχαντιστές που δολοφονούν στο όνομα του Ισλάμ. Οι μειονότητες είναι πλέον εγκλωβισμένες μεταξύ ενό καθεστώτος που δεν τις προστατεύει πλέον αλλά καταδιώκει και ταυτόχρονα με τους τζιχαντιστές που θέλουν να ε, έχουν ε, θρησκευτικά αντίπεινα και όπου μπορούν να οργανώσουν κοινέ επιχειρήσεις με κατά του τοπικού πληθυσμού. Εδώ λοιπόν τα δίκτυα αυτά, τα τρομοκρατικά δίκτυα που υποφελούνται από το χάο του πολέμου θα ε, ριζώσουν στην περιοχή αυτή απειλώντα ολόκληρη τη γεωγραφική ζώνη αλλά και την Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Γιατί υπάρχει χρηματοδότηση για αυτέ τι ομάδε και αυτό πρέπει να μα απασχολήσει. όλε οι που φέρουν διπλά από τον πόλεμο ω πολίτες αλλά και ω ε, στόχοι ε, θρησκευτικών και εθνοτικών επιθέσεων. Είναι λοιπόν καθήκον μα, αλλά και καθήκον τη Συριακή κυβέρνηση και ολόκληρη ολόκληρη τη ε, διεθνού κοινότητα να προστατεύσουμε τι ευάλωτε αυτέ ομάδε. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου μου που βρίσκονται εδώ σήμερα ε, πέμπτη απόγευμα για να ε, βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο τη Συνόδου Ολομέλεια, όπου υπάρχει σύγκληση απόψεων μετά των πολιτικών ομάδων. Και ευχαριστώ και τον κύριο Πόσελτ, τον οποίο περίμενα να συμμετάσχει μαζί μας. Ευχαριστώ. Σάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Είναι απίστευτο ότι ε, τελειώνουμε την σύνοδο αυτή με ψήφισμα για τη Συρία. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα. Και έχουμε μια τεράστια αντίθεση μεταξύ της, των φρικαλωτήτων επιτόπου και της, ε, της άδειας ολομέλειας σε όλες τις ε, συζητήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι πραγματικά ένα γερτήριο για όλους μας. Ε, θα πρέπει να θυμηθούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω από 150.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν εσωτερικά. 2,5 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες βρίσκονται σε γειτονικέ χώρες και δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για αυτό τον ε, αποτρόπαιο πόλεμο. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε επιτέλου, Σήμερα επικεντρωνόμαστε στι μειονότητε και στην ιδιαίτερα ευάλωτη θέση του. Εθνοτικέ και θρησκευτικέ μειονότητε, αλλά και γυναίκε και παιδιά που υποφέρουν δυσανάλογα μεταξύ των αμάχων και βρίσκονται στα διασταυρούμενα πυρά μεταξύ εξτρεμιστών τζιχαντιστών και ένα δολοφονικό καθεστώ. Θα ήθελα να απευθύνω από τι από τη στον Πάτερ Βαντερλούχτ που έχασε τη ζωή τον Απρίλιο. Ε, γιατί ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι εξακολουθούν να είναι θύματα αυτής της κρίσης. Ακόμη και η Ραζάν Ζαϊτουνέχ, βραβείο Ζαχάραβ 2011, απήχθη με το σύζυγό της και δύο άλλους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από τέσσερις μήνες ε, και θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση για την απελευθέρωσή της. Το καθεστώς Ασάντ χρησιμοποιήσει την θρησκευτική πόλωση ως στρατηγική επιβίωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να μην πέσουμε και εμείς στην παγίδα εντείνοντας τις διαφορές ε, και να ε, εξωθήσουμε μία μειονότητα έναντι άλλης. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων συνδέονται άρρηκτα με το σεβασμό και άλλων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότητα, καθώς και το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Μία λύση μετά από διαπραγμάτευση θα απαιτήσει υποχωρήσει και συμμετοχή και από το Ιράν, τα κράτη του κόλπου και τη Ρωσία. Και θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κοινωνία που όλοι οι Σύριοι θα μπορούν να διαβιούν ελεύθερα. Αλλά έχουμε δυστυχώ πολύ μακρύ δρόμο να διανύσουμε για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, κυρία Σόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικότητα ότι έχουμε ήδη ψηφίσει αρκετά ψηφίσματα για τη Συρία το τελευταίο χρόνο, αλλά είναι προφανές ότι το να μιλάμε για ευάλωτες κοινότητες δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε όλους τους πολίτες της Συρίας από την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόνται αυτή τη στιγμή. Πράγματι είναι εκατομμύρια τα άτομα που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή στη Συρία. Είναι περίπου 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στις γειτονικές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να θίξω δύο ε, διαστάσεις του θέματος. Ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα από ό,τι θα έχει κάνει ως τώρα και ότι επίσης πρέπει να μιλάμε για τον πληθυσμό των Κούρδων και των ε, Παλαιστινίων. Διότι δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπε ε, ομάδε πληθυσμού στην ε, Συρία δεν χρήζουν τη ε, ίδια προστασία, αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητε για του Κούρδου καταρχήν. Για του Κούρδου, οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα με το Ιράκ και την Τουρκία και υπάρχει εμπάργκο για την ανθρωπιστική βοήθεια στι περιοχέ αυτέ. Οπότε πλήττονται. Επίση, η διαδικασία εκδημοκρατισμού τη Συρία θα πρέπει να λάβει υπόψη τι ιδιαιτερότητε όλων των πληθυσμών που βρίσκονται στη χώρα. Το ίδιο και για τον πληθυσμό των Παλαιστινίων. Να θυμίσω ότι υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ε, προσφύγων από την Παλαιστίνη που βρίσκονταν ήδη στη Συρία ως πρόσφυγες και τώρα θα πρέπει να φύγουν και από εκεί και να πάνε στις γειτονικέ χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να θυμίσω ότι επειδή ο Λίβανος είναι μια χώρα πάρα πολύ μικρή και έχει ήδη υποδεχθεί ένα μεγάλο αριθμό Σύρων προσφύγων εκ των οποίων ένα, μέλος, ένα μέρος μόνο ήταν Παλαιστίνοι θα πρέπει ε, και εκεί να σκεφτούμε την αποστολή ανθρωπιστική βοήθεια. γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει ούτε ευρωπαϊκή βοήθεια ούτε τίποτε άλλο. Και αυτό γιατί δεν υπήρξε πολιτική βούληση. Αλλά και γιατί υπήρξαν και άλλες περιπλοκές ε, και επιπλοκέ πολιτικού χαρακτήρα εκεί. Επίσης, στον καταπλησμό Άρμο που είναι ένα καταπλησμός προσφύγων, Παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία. Εκεί ε, οι διαφιλονικίες μεταξύ αντιπολίτευσης και του πολιορκίες τη κυβέρνηση δεν επέτρεψαν να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Σόζα. Ευχαριστώ κυρία Φλότρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε δεν έχουμε πια στη Συρία κοινότητες που δεν είναι πια ευάλωτες. Από τότε που ο Ασάντ και το καθεστώς του αποφάσισε με κάθε μέσο να εξολοθρεύσει τις εύλογες δημοκρατικές προσδοκίες του λαού του. Όλες οι κοινότητες, όλες οι ομάδες πληθυσμού είναι σήμερα υπό απειλή στη Συρία. Πρόκειται για ένα σπιράλ βίας ανήκουστο, απίστευτο, χωρίς όρια. 150.000 θάνατοι, 6.500 εσωτερικά εκτοπιστέντες, 2.500 πρόσφυγες ε, εκτός Συρίας. Ε, έχει πολλές τεχνικές πολεμικές ο Ασάντ. Ε, στρέφεται κατά σχολείων, ε, ε, νοσοκομείων, συναθρήσεων, καταστήλει και καταπιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και χημικά όπλα χρησιμοποιεί. Έχουμε ε, ε, μαζικές επιθέσεις με, TNT, με βαρέλια TNT με νητρογλυκερίνη στρέφεται κατά του πιο ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού των αμάχων. Το είδαμε αυτό στο Χαλέπι. Και επίσης ε, έχουμε ε, τεκμήρια για συστηματική και μαζική χρήση των βασανιστήριων ως ε, εργαλείου πολέμου. Το καθεστώς Ασάντ είναι μηχανισμός δολοφονίας ουσιαστικά και αυτή η βαναυσότητα του πολέμου απειλεί σήμερα όλες τις κοινότητες ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και απειλή εξαιτία τη ε, αύξηση των θρησκευτικών, εξτρεμιστικών, τζιχαντιστικών, ε, παραστρατιωτικών, ε, φιλοκυβερνητικών ή αντικαθιστωτικών ομάδων. Είναι άπειρε οι τέτοιε ομάδε που πολλαπλασιάζονται. Έχουμε Ασσυρίου, Άραβε, Κυρκασίου, Κούρδου, Τουρκμένου, Αραμαίου, Αρμενίου, Αλαουίτε, μουσουλμάνους, Σουνίτες, χριστιανούς, δρούζους, όλοι αυτοί δεν πρόκειται να τύχουν ε, ε, προστασίας αν δεν αποκατασταθεί η δημοκρατία και η ελευθερία στη Συρία και ε, μια κυβέρνηση που θα σέβεται τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Τι μπορεί να κάνει σήμερα η Ευρώπη. Η μόνη της επιλογή είναι να να ενισχύσει πάση θυσία τη δημοκρατική αντιπολίτευση παρά τις δυναμίες της που δέχεται τη διαπραγμάτευση και κάνει ό,τι μπορεί. Διακόπτεται δυστυχώς το μικρόφωνο της κυρίας Φλότρ. Σας ευχαριστώ. Ε, ο μιλητής ξενόμου των ομάδων. Ε, κυρία Σαγιαή ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε συνεχώς για την Ουκρανία, αλλά καλό είναι να σκεφτούμε λίγο και το τι γίνεται στη Συρία. Πάρα πολλοί χριστιανοί σε ολόκληρο τον ε, κόσμο σήμερα πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά στην ε, Συρία υποφέρουν από διώξεις, όπως είπαν ε, και οι συνάδελφοι. Το θέμα αφορά όλες τις μειονότητες. Η Human Rights Watch έγραψε μία έκθεση ειδικά για το τι γίνεται εμποδίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε στρατόπεδα προσφύγων. Ε, στο Σαλάμ κοντά στην Τουρκία υπάρχουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι και δεν αφήνουν να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια γιατί δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Ρέπο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καταστροφή αυτή, η σύγκρουση αυτή οδήγησε μια ανθρωπιστική καταστροφή που δεν έχουμε δει. Ο Συριακός λαός αποτελείται από πολλές ε, εθνικές ε, και θρησκευτικές κοινότητες. Κινδυνεύουν κυρίως οι θρησκευτικές μειονότητες. Η Συρία μέσα από την ποικιλομορφία κατέληξε να είναι ένα σύμβολο ε, σύνολο με συγχωρείτε διαφόρων μειονοτήτων ένας εθνικός πλούτος που πρέπει να προστατευτεί. Οι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες έχουν την ευθύνη να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει πως τα λόγια της σημαίνουν κάτι. Γιατί λόγια, λόγια, λόγια και από πράξεις τίποτα. Πρέπει να γίνει κάτι. Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, τουλάχιστον κάτι με τους προσφύγεις. Ευχαριστώ. Μπιλμπάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. 150.000 θύματα έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπιστέντες. Πάνω από 2,6 εκατομμύρια πρόσφυγες. Θηνωτικές και θρησκευτικέ μειονότητες βρίσκονται υπό ιδιαίτερη απειλή. Πάνω από 540.000 Παλαιστίνοι πρόσφυγες μεγάλος αριθμός προσφύγων ε, γυναικών και παιδιών που υφίστανται σεξουαλική βία και επιθέσεις. Τρία εκατομμύρια παιδιά κατέληψαν το σχολείο από το 2011 και πάνω από 500.000 δεν έχουν εγγραφεί στα σχολεία. Θρησκευτικέ δολοφονίες, απαγωγές. Αυτή είναι η φωτογραφία. Αυτό είναι το στιγμιότυπο της Συρίας και δυστυχώ το μόνο που κάνουμε είναι να, κατηγορούμε του εξτρεμιστέ και το καθεστώς Ασάντ. Έχουμε κατάφορη παραβίαση του, ε, του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια διαπραγμάτευση, να προστατεύσουμε τις μειονότητες που δεν έχουν πόρους, να προσαχθούν σε δικαιοσύνη δράστες των εγκλημάτων. Θα πρέπει να επέβουμε με πολιτικό τρόπο για να αποτρέψουμε τις καταστροφές. Ο λόγος, ο διάλογος και η αποδοχή της πολυμορφίας είναι το καλύτερο αντίδοτο κατά των τεθωρακισμένων του καθεστώτος. Ε, θα ήθελα να επιθυμίσω και ένα άλλο δράμα, την εγκατάλειψη, την ε, ε, εξαφάνιση ενός Βάσκου στην Αμβέρσα. Και συνεχίζει στα βασικά η κυρία Μπαραντίκα. Δεν εσπεράντσας. Μιέσκερ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Κλούτε. είναι νομίζω σημαντικό το ότι αναφερθήκαμε στην Συρία όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, πράγματι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Η κατάσταση είναι δραματική, αλλά θα ήθελα να επιθυμίσω εδώ πως υπάρχουν και κάποια σημεία ελπίδας. Οι κουρδικές περιοχές στο βορρά μέχρι στιγμής κατάφεραν να ξεφύγουν από τη βία και να φτιάξουν κάποιες βασικές δημοκρατικές δομές. Πάνω από ένα εκατομμύριο Σύριοι άρα έχουν καταφύγει σε αυτές τις περιοχές, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αλλά η περιοχή αυτή απομονώνεται από τους γείτονε και από την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τη στάση της Τουρκίας εάν είναι, να, ε, είναι υποψήφια χώρα. Πρέπει επιτέλους να ανοίξει τα σύνορά της εκεί πέρα, να αφήσει να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και απευθύνω εδώ πέρα έκκληση στην τουρκική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Γκρίφιν για ένα λεπτό. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε. Το δράμα των μειονοτήτων και των προσφύγων στη Συρία είναι φοβερό, αλλά από ποιον προσπαθούν να αποδράσουν. Πήγα δύο φορέ στην Συρία το περασμένο καλοκαίρι και με επιστολέ προ τη Συριακή κυβέρνηση προσπάθησα να μιλήσω για, τις, για του βομβαρδισμού που δεν θα έπρεπε να πλήττουν τη Συρία με τη στήριξη τη Βρετανική κυβέρνηση για την προστασία των χριστιανών και μουσουλμάνων προσφύγων. Να σα πω όμω ότι τεράστιο αριθμό του έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια του, από τι αιστείε του, από του ίδιου τζιχαντιστέ του οποίου αθελάτε βοήθησε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να βοηθήσουμε τη Συρία, θα πρέπει η CIA και οι τζιχαντιστέ να σταματήσουν να οπλίζονται ε, και να οπλίζονται μισθοφόροι του. Θα πρέπει να επιφληθούν κυρώσει στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που έχουν ε, ε, ουσιαστικά χρηματοδοτήσει την εισβολή στη Συρία των, κατά των χριστιανών και των σουνιστών που προσπαθούν να υπερασπιστούν τη ζωή του. Ευχαριστώ κύριε Γκρίφιν. Στάσνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, είμαι ενθουσιαδός υπέρ του ψηφίσματος ε, και υποστηρίζω όλες τις προσπάθειες τη διεθνής κοινότητας ε, να εξεύρουν λύσεις για να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στη Συρία εκατομμύρια αθώοι έγιναν θύματα. 12.000 άνθρωποι φεύγουν από τη Συρία κάθε εβδομάδα και ήδη 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τη Συρία, ενώ 3,5 έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. Αυτή η ανθρωπιστική κρίση είναι πραγματικά πρωτοφανής. Είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες ε, του, της σύγχρονης εποχής και μάλιστα θύματα είναι όλοι και κυρίως αθώοι, άμαχοι ή μέλη θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, οι χριστιανοί για παράδειγμα. Για να επιληθεί η κατάσταση θα πρέπει να βρεθεί μία λύση δημοκρατική, ειρηνική, με τη Συρία να πρωτοστατεί και την διεθνή κοινότητα να υποστηρίζει θα πρέπει να βρεθούν οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων και από τις δύο πλευρές αυτής της αίματηρης σύραξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σένισιν. Ευχαριστώ. Ε, στυλιτεύουμε απερίφραστα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην Συρία, ιδιαίτερα των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων. Η Συρία είναι πολύ όμορφη χώρα από θρησκευτική και εθνοτική άποψη, γι' αυτό και η αναζήτηση αποτελεσματική ε, ε, πολιτικής λύσης ε, προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Ένα νέο πολιτικό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσει ίσα δικαιώματα άσχετα από την προέλευση και την καταγωγή, την ομολογία, τη δοξασία ή τις πεπιθήσεις και τη θρησκεία. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη την ε, πολυμορφία της ε, συριακής κοινωνίας και επίσης θα πρέπει να είμαστε αυστηρά υπέρ τη στηρίσης του δικαίου και να, να στυλιτεύσουμε την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών και την στρατολόγηση ανηλίκων. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της Συρίας. Πολύ συχνά ε, απευθύναμε έκκληση να διορθωθεί η κατάσταση στη Συρία και επίσης να επιληθεί και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την δίωξη των εγκλημάτων. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Και εδώ πέρα ε, έχουμε πάλι διπλάσιους που έχουν ζητήσει το λόγο διπλάσιο από το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Ο κύριος Ζιμπ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όλε οι μέχρι τώρα προσπάθειες για την, για την ε, άμβληση της κρίσης στη Συρία δυστυχώς ήταν αναποτελεσματικές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση. Ενώ ε, ο μισός πληθυσμός της Συρίας έχει εκτοπιστεί εσωτερικά. Έχουμε πάνω από 150.000 θύματα που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία απαιτούν άμεση αντίδραση της παγκόσμιας κοινότητας. Διώκονται κυρίως μέλη μειονοτήτων, ε, για παράδειγμα χριστιανοί. Επίσης, ε, θα πρέπει ε, ταυτόχρονα με λύση της ε, σύραξης να ζητήσουμε και προστασία των μειονοτήτων. Γιατί τελείως δεν νοείται ε, ειρηνική λύση. Για παράδειγμα, έχουμε Αραμαίους στη Συρία. 2.500 άνθρωποι μιλούν την αραμαϊκή στη Συρία. Είχαμε την περίπτωση στην πόλη Μαλούλα. Δραματική κατάσταση των, της αραμαϊκής κοινότητας. Η αραμαϊκή γλώσσα που είναι η γλώσσα από την εποχή του Χριστού και την μιλούν 2.500 άνθρωποι δυστυχώς ε, δεν ε, ακούγεται. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τέτοιες μειονότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σέγγεντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συναδελφοί λυπούμε για το τι έχουμε κάνει σε σχέση με τη Συρία δεν είμαστε καν πιστοί στα δικά μας ιδανικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι δεν είναι μόνο συσσωμάτωση των κρατών μελών, αλλά προστατεύει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζω πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δραματική. Υπάρχουν ε, χιλιάδες νεκροί, συγκρούσεις, τυχές ε, με τις μονάδες της, ε, κινδυνεύει η ειρήνη, κινδυνεύουν οι θρησκευτικές ε, μειονότητες. Γι' αυτό πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιηθεί περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ δεν θα ξανακάτεβω στις εκλογές, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω εσά που θα συνεχίσετε να προστατεύετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο κύριο Σόνικ. Ε, από του υπόλοιπου ζητώ κατανόηση. Ευχαριστώ. Του τελευταίου μήνε παρατηρούμε αυξανόμενη δράση των ε, Ισλαμιστών εξτρεμιστών. Έχουμε όλο και περισσότερε επιθέσει ε, κατά μελών ε, θρησκευτικών μειονοτήτων στη Σύρια. Επίσης έχουμε πολλές ε, βίες, πράξεις και βαναυσότητες ε, σεξουαλικού χαρακτήρα κατά γυναικών και παιδιών, καθώς και επιθέσεις κατά ακτιβιστών, ιερωμένων ε, ή δημοσιογράφων. Η Συρία θα πρέπει να τηρήσει και το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να επέμβουμε άμεσα εκεί για να σταματήσουν επιτέλου αυτέ οι καταστολέ και οι επιθέσει. Επίση, θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή της, των Συριακών Αρχών αλλά και τη παγκόσμια κοινότητα στην κλιμάκωση αυτή τη βία, Γιατί αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμό των θυμάτων, κάτι που δείχνει ότι η σύραξη δεν αφορά μόνο πολιτική διαμάχη αλλά και εθνοτική και θρησκευτική αντιπαράθεση με αποτέλεσμα να υποφέρουν πάρα πολύ αθώοι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρωθήκε η διαδικασία. Τον λόγο έχει ο κύριος Αλμούνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το κατεπήγον ψήφισμα για την κατάσταση στην Συρία. Ιδίω για να υποστηρίξει τις πλέον ευάλωτες κοινότητες στη χώρα αυτή. Η κατάσταση στη Συρία συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ανησυχητική, με ένα δύο εμφύλιο πόλεμο εξέλιξη. Η, Ευρω... η διεθνής κοινότητα έχει προσπαθήσει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στην Γενέβη σε μια δεύτερη φάση αλλά όλα αυτά διακόπηκαν λόγω τη επανεκλογή του πρόεδρου Ασάντ. Το Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτέ τι εκλογέ και είπε ότι θα ήταν μια παροδία για οποιαδήποτε δημοκρατική προσπάθεια κάτι τέτοιο, χωρί καμία εξοπιστία. Όμως είχαμε τοπικός και τη βίαιη ε, καταστολή από το ε, καθεστώς του Ασάντ που έχει προσελκύσει και τρομοκρατικές ομάδες με επιθέσεις κατά των πλέον ευάλωτων και αθώων όπως με την ε, επίθεση κατά της πόλης ε, Κασάτ. Η, η ύπατη εκπρόσωπο Άστον έχει καλέσει τους αγωνιστές αυτές να εγκαταλείψουν την Συρία και τους εξωτερικούς τους υποστηρικτές να πάψουν να τους υποστηρίζουν. Το καθεστώς έτσι κι αλλιώς υπολογίζει στην εξωτερική αυτή υποστήριξη που επιδεινώνει την κατάσταση και δεν επιτρέπει να βρεθεί μια λύση εκ των έσω στην περίπτωση της Συρίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με όλους τους ενδιαφερομένους προκειμένου να να διατηρηθεί η προσπάθεια πολιτικής εξέβρεση πολιτική λύση. Όμω δυστυχώ η κατάσταση για τους χειρούς επιδεινώνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί σε όλα τα μέτωπα να υποστηρίξει τον πληθυσμό τη χώρα αυτή και έχει δείξει τον πρωταγωνιστικό τη ρόλο στη διεθνή κοινότητα Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθεια, πιέζοντα για να υπάρξει πρόσβαση, δυνατότητα αποστολής τη βοήθεια αυτή με το πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ 2139 προκειμένου να υποστηριχθούν οι πρόσφυγες ε, όλων των υπόλοιπων εθνικών κοινοτήτων όπως οι ε, Παλαιστίνοι αλλά και οι χώρες υποδοχής των προσφύγων και να μπορέσουν βεβαίως οι Σύριοι να ξαναοργανώσουν τη ζωή τους σε όλους τους τομείς. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις δραστηριότητες υποστήριξης των πλέον ευάλωτων, τους πρόσφυγες, τους εσωτερικώς εκτοπισμένους, τους πολυερκημένους, τις γυναίκες και τα παιδιά, τις μειονότητες μεταξύ των οποίων χριστιανούς και στο, Υπουργείο στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων την Δευτέρα ε, επαναβεβαιώθηκαν οι στόχοι αυτοί. Η υπάτη εκπρόσωπο Άστον εξέφρασε την ε, αποτροπή της για την δολοφονία του πατρός Φαντελούχτ έναν τον άνθρωπο που βοήθησε τόσους ε, Σύρους πολίτες στην πόλη της Χόμς. Και άλλοι όμως ακτιβιτές, οι, οι Ρωμένοι συνεχίζουν να πάγονται. Ε, κυρίω από εξτρεμιστικέ ομάδε ή ομάδε που έχουν διασυνδέσει με την Αλκάιντα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ζητά τη λογοδοσία ώστε να βρεθούν οι δράστε αυτών των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα και των παραβατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του διεθνού δικαίου, γιατί όσοι έχουν γίνει κατά των πλέον ευάλωτων δεν θα περάσουν έτσι. Ευχαριστώ. Κύριε Αλμούνια. Εφτά ψηφίσματα έχουν κατατεθεί. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλο τη επόμενη συζήτηση. Επόμενο θέμα. Η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Ο κύριος Μπίελεν για δύο λεπτά.